Καλό σας απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε λοιπόν την απογευματινή μας ημερήσια διάταξη, αλλά πρώτα απ' όλα να συζητήσουμε τα πρακτικά και τα κείμενα της, χετινής, της χθεσινής συνόδου. Τα έχετε λάβει και αν δεν υπάρχουν σχόλια θεωρούνται ως συγκεκριμένα τα πρακτικά. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Περνώντα το πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξη. έχουμε τρία σχέδια ψηφίσματος για την Ικαράγουα και θα δώσω το λόγο στους ε, εισηγητές. Συντάκτε των ψηφισμάτων. Πρώτος ο κύριος Μπογκούσο Αφασόνικ. Πολιτικά. Ευχαριστώ. Η πολιτική του Δανιέλ Ορτέγκη, του ισχύοντος του ενεργεία προέδρου της Νικαράγουας, είναι η νοοτροπία της παλιάς κομμουνιστικής ε, ιδεολογίας από τη στιγμή που, κρατάμε, που λαμβάνουμε την εξουσία δεν την αφήνουμε από τα χέρια μας και μετά την, τους αντινίστες η Νικαράγουα χρειάστηκε να αποδεχθεί τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού και μάλιστα το 2006 ε, ο Ορτέγα επανήλθε στην εξουσία, οι σαντινίστες ανέλαβαν και πάλι τα ενία και άρχισαν ε, με ψευδονομικίστικους ε, στόχους να προσπαθούν να εξαλείψουν την αντιπολίτευση. Και μάλιστα κυριάρχησαν σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας. Μάλιστα πριν από λίγα χρόνια εμείς ε,